Το λόγο έχει ο συντάκτης κύριος Λάγκε για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι όλοι μας ε, Έχουμε, είμαστε ακόμα αγανακτισμένοι με αυτά που συνέβησαν στον Μπαγκλατές, ε, το ατύχημα αυτό στον Μπαγκλατές, αλλά και πάρα πολλά άλλα ατυχήματα όπου οι άνθρωποι όπου πάρα πολλοί άλλοι ε, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη σωματική τους ακερότητα. Γι' αυτό λοιπόν έκρινα ότι ήταν απολύτως απαραίτητο μετά το ατύχημα στη Ράνα Πλάζα να οργανωθούμε και να συζητήσουμε για το σύμφωνο της βιωσιμότητας το οποίο ε, συνοδεύεται από μια συμφωνία για την παραγωγή και για το ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που να ισχύουν στον Μπαγκλαντές. Αύριο λοιπόν θα ακολουθήσει η τρίτη συνάντηση και ελπίζω όλα αυτά να στεφτούν από επιτυχία. Θα είναι βέβαια επιτυχία μόνο αν επιτευχθεί και μια σαφής ε, συμφωνία για το πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση. Γι' αυτόν λοιπόν το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Αμφίβολα έχουν υπάρξει έχει υπάρξει πρόοδος, ε, έχουμε μία αλλαγή του νόμου ε, του εργασιακού, έχουν συστηθεί καινούργια συνδικάτα και κυρίως όσον αφορά τους μισθούς ε, και τις ε, συνθήκες ε, εργασίες. Οι δυνατότητες της συλλογικής δράσης είναι καθοριστική σημασία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε βελτιώσεις. Επίσης, επιτύχαμε, είδαμε ότι υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού και μόνο αυτό αλλά σε, χίλιες σε 1700 εργοστάσια στο Μπαγκλατές έχουν υπάρξει ε, επιθεωρήσεις ε, για την ασφάλεια του κτηρίου αλλά και για την ε, πυρασφάλεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι επιτύχαμε αρκετά πράγματα. Βεβαίως ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας μας προειδοποιεί και μας επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Ε, είμαστε πολύ τυχεροί για το ότι η Κομισιόν το αναφέρει αυτό σε μια δική της επιστολή. Κατόπιν τούτου, κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι δυνατόν από τη μία πλευρά στο Μπαγκλαντές το ίδιο το Μπαγκλαντές να χρησιμοποιεί και με αποτελεσματικότητα μάλιστα το θέμα των τιμών γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια το Μπαγκλαντές έχει επιτυχεί και μία ανάπτυξη της τάσης ε, της τάξης του 6,6%. Όσον αφορά όμως ε, την αναγνώριση των δικαιωμάτων εργαζομένων Εκεί δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις. Υπάρχει λοιπόν ένα ψήφισμα για την κλωστεφαντουργία, θεσπίστηκε στην προηγούμενη Ολομέλεια και εκεί αναφέρουμε ότι θα πρέπει να ισχύουν δεσμευτικοί κανόνες για την τήρηση των ε, κριτηρίων βιωσιμότητας ακριβώς όπως προβλέπεται στις οδηγίες του ΟΣΑ. Και μόνο αυτό, αλλά το προτιμησιακό μας σύστημα θα πρέπει να το προσαρμόζουμε περισσότερο ε, στην τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν ε, στο πλαίσιο του ΕΛΙΤΣΙΣ να τα δεχόμαστε όλα και σε τελική ανάλυση και το Μπαγκλαντές θα πρέπει να εξάγει τα δικά του τα συμπεράσματα. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τι ακριβώς γίνεται ε, με τα δικαιώματα εργαζομένων στις ε, ειδικέ ζώνες εξαγωγών. Υπάρχει μια συμφωνία και με βάση αυτήν η κυβέρνηση υποτίθεται θα αναθεωρήσει τις σχετικές διατάξεις, αλλά χρειαζόμαστε ε, σαφήνεια. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο κατηγορίες εργαζομένων. Ε, το σύστημα καταγραφής των συνδικάτων και επίσης και το θέμα της εργασίας ε, στα εργοστάσια, όπως επίσης και το θέμα της που ασκείται έναντι των συνδικάτων, όλα αυτά δεν είναι αποδεκτά. Ως εκ τούτου, ε, το εξή ερώτημα για μας. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ε, να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Διεθνούς ε, οργανισμού Εργασίας και πάνω απ' όλα θα πρέπει να παρατείνουμε τη συμφωνία και μετά το 2018 γιατί δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει το έργο μας. Αυτή είναι η ερώτηση που απευθύνουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Λάγκη. Καλησπέρα σε όλους. Η κυρία Μάλστρομ, ε, εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που βάλατε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας για το σύμφωνο και τις ανησυχίες σας για τον Μπαγκλαντές. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν είναι δεσμευμένη να αντιμετωπίσει τα πρότυπα εργασίας και στην, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής. Έχουμε τις συμφωνίες ε, εμπορίου και επενδύσεων, έχουμε τις ε, συμφωνίες, ε, τις ειδικές, έχουμε το σύμφωνο βιωσιμότητας και έχουμε και τα, τις ειδικές προτιμήσεις, το SPG. Λοιπόν, ο Διεθνή Οργανισμό Εργασία έχει μια ειδική παράγραφο για τον Παγκλητέ στην περσινή έκθεση για, για τι λογικέ συμβάσει και για την ελευθερία ε, του συνέρχεστε. Είναι σοβαρή προειδοποίηση. Επίση, ε, οι ευρωβουλευτέ, κάποιοι ευρωβουλευτέ, ε, επισκέφτηκαν τον Παγκλητέ και το μήνυμα που στείλατε είναι πάρα πολύ δυνατό και βάζει πραγματικά το θέμα φωτίζει το θέμα, το βάζει στην ημερήσια διάταξη, δημιούργησε έτσι μια συνειδητοποίηση για τα προβλήματα και ε, χάρη σε αυτέ τι προσπάθειε, ε, κάπω κινητοποιήθηκε η κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ. Φυσικά, συμφωνώ με το στόχο ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ θα πρέπει να σέβεται πλήρω ε, τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Τώρα, για τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτετε, κύριε Λάγκε, και οι υπόλοιποι. Ε, υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια από το Μπαγκλατέ σε εργασιακό μέτρο. Υπάρχουν τριμερεί συμφωνίε από το Φεβρουάριο Φέτο και Επίσης υπάρχουν οι νόμοι για τις ε, ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών που δεν ε, συνάδουν με το ILO και που τις έχουν αναστείλει. Ε, αυτές οι τριμερείς διάλογος είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να αναθεωρήσει όλο το εργασιακό δίκαιο και αυτό είναι θετικό σημάδι. Θα πρέπει να το καλωσορίσουμε και να το αναγνωρίσουμε παράλληλα. γίνονται, ακούγονται ερωτηματικά για την παράταση της εντολής ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε και μετά το 2018, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να βελτιώσουμε περαιτέρω τα πράγματα. Χρειάζεται να γίνει σοβαρή προσπάθεια γι' αυτό. Τι θα κάνουμε αύριο. Όπως είπε ο κύριος Λάγκη, θα έχουμε τη συνάντηση follow-up της ε, ομάδας για το υψηλό επίπεδο για το σύμφωνο βιωσιμότητας η οποία θα καταγράψει το που έχουμε φτάσει και θα συζητήσει το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Έχουμε ξεκαθαρίσει στις αρχές του Μαγκλαντές ότι περιμένουμε να αναλάβουν ε, κατεπηγόντως δράση σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μια νυχτή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, σαφής, διαφανή, διαφανής ε, με συγκεκριμένα ορόσημα. Ε, θα πρέπει να δούμε τις λογικές συμβάσεις εκεί και την ελευθερία του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε. Θα πρέπει να καταχωρούνται γρήγορα τα συνδικάδα τα συνδικάτα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν και έρευνες και διώξεις όλων των ε, δράσεων ε, που, είναι, που συνιστούν διάκριση ή κατά των συνδικάτων. Επίσης θα πρέπει να θεωρηθεί το, ο νόμος ε, για τα εργασιακά θέματα του μπαγκλατέ, καθώς και ο νόμος για τις ελεύθερες μηχανικές ζώνες εξαγωγών και να σέβεται τα όσα επιτάσσει ο ILO. Επίσης, θα πρέπει ε, να υπάρχει μια εντολή και αναθεώρηση της εντολής ε, της συμφωνίας. Θα πρέπει να βρούμε και τρόπους να διευκολύνουμε το διάλογο μεταξύ διαφόρων ε, ε εμπορικών σημάτων και των ε, υπεργολάβων τους. Θα πρέπει να υπάρχουν τεχνικά εργαστήρια, συνεργασία με τον ΩΣΑ για θέματα ετοίμων ενθυμάτων με ειδική εστίαση στις πρακτικές αγοράς θα πρέπει να υπάρχουν ε, διεθνείς φορείς στους οποίους θα βασιστούμε ε, θα πρέπει να ε, βασιστούμε όπως ας πούμε στον εξειδικευμένο φορέα που αποτελεί το ILO. Το σύμφωνο, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σημαντικό πλαίσιο για να συζητήσουμε τον Παγκλατέ και μαζί με άλλου διεθνού εταίρου για τα εργασιακά δικαιώματα. Εάν δεν υπάρξει επαρκή πρόοδο σε εύλογο χρονικό διάστημα, η Κομισιόν θα πρέπει να δει τι άλλε δράσει μπορεί να προωθήσει. Έχουμε εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο κανονισμός JSP και ξέρετε ότι ο κανονισμός αυτός προβλέπει ε, προσωρινή απόσυρση των ε, εμπορικών προτιμήσεων σε περίπτωση σοβαρής και συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό είναι εργαλείο. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος στο, από πλευράς Μπαγκλαντές και ελπίζω ότι η αυριανή συνεδρίαση θα οδηγήσει σε κάποια πρόοδο, αλλά εμείς θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης της εξελίξης. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το ενδιαφέρον σας, για τη συμμετοχή σας. Ε, καλό είναι να συνεργαστούμε και να στείλουμε και οι δύο το ίδιο ε, ηχηρό μήνυμα στις αρχές του Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα ας ακούσουμε τους πολιτικές ομάδες από το ΕΛΚ, ο κύριος Ρούας, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Καρίμ για τα όσα έκανε σχετικά με το σύμφωνο βιωσιμότητας που υπεγράφει το 2013 μετά το τραγικό ατύχημα στο Ραν Πλάζα. Το 2013 επαναλαμβάνω. Να μην ξεχνούμε ότι έχασαν τη ζωή τους το 2013 1.100 άνθρωποι. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξανασυμβεί παρόμοια τραγωδία. Το θέμα παραμένει δυστυχώς εξαιρετικά επίκαιρο, ενώ βεβαίω τη συναντήση αύριο στην ΤΑΚΑ. Κύριε Επίτροπε, θέλω να ζητήσω μέσω ημών από την Επιτροπή, εν το σύνολο τη, να μην ξεχάσουν τον Μπαγκλαντές. Δεν πρέπει να διστάσουμε ούτε λεπτό. Να ασκήσουμε περαιτέρω πίεση στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Ταυτόχρονα ο, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας και ο ιδιωτικός τομέα συνεχίζουν να πιέζουν για να πετύχουν αυξημένη συμμόρφωση στον συγκεκριμένο τομέα, στην εφαρμογή δηλαδή του Συμφώνου Βιωσιμότητας. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος βεβαίως στις συνθήκες εργασίας κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια στα κτίρια και βεβαίως ε, θα συγχαρώ ως προς αυτό τις αρχές του Μπαγκλαντές. Όμως η συνεχιζόμενη πρόοδος πρέπει να επαληθευθεί και να επαληθεύεται διαρκώς. Γιατί τώρα τελευταία προς τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν είδαμε κάτι. Πρέπει να τροποποιηθεί και η εργασιακή νομοθεσία. Ε, στον τομέα, για παράδειγμα, της ε, ελευθερίας του συνεταιρίζεστε στον κανονισμό 87-98 όσον αφορά το κράτος δικαίου, την διαφθορά, τις προληπτικές αυθαίρετες συλλήψεις, τις ε, έρευνες και ανακρίσεις και ούτω Τέλος, θυμίζω ότι η νομοθεσία που διέπευθε στις ελεύθερες ζώνες πρέπει να συμμορφωθεί με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα γιατί οι καταχρήσει συνεχίζονται ακόμη. Ευχαριστώ. Από τους, από 1,5 λεπτό για τον κύριο Γιονγκέριου, Κυρία Γιονγκέριου. Ευχαριστώ. Τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το σύμφωνο βιωσιμότητα και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι εργασιακέ συνθήκε των Μπαγκλαντές είναι αρκετά κακέ ακόμα και σε μερικέ περιπτώσει, παραδείγματο χάρη τα δικαιώματα των συνδικάτων, ε, είναι και χειρότερε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευτυχώ το αναγνωρίζει αυτό και η επιστολή που εστάλει στον πρέσβη του Μπαγκλαντές στις Βρυξέλλες από τη Γενική Διεύθυνση ΕΜΠΛΕ, ΔΕΒΕ και Εμπορίου προειδοποίησε τη χώρα ότι έχουν μέχρι τις 18 Μαΐου για να σημειώσουν επαρκή και ουσιαστική πρόοδο καθώς και να ετοιμάσουν μια ουσιαστική στατηγική ε, για να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα της, της εργασιακής νομοθεσίας. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει μια ε, έρευνα στα πλαίσια του GSP, του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων. Η 18η Μαΐου είναι αύριο και ξέρετε πολύ καλά ότι ε, έχει ακυρώσει αυτού τους εργασιακούς νόμους το Μπαγκλαντές, αλλά δεν έχουν γίνει άλλες ουσιαστικές κινήσεις. Φυσικά, Έχουμε ακόμα μερικέ ώρες μέχρι τις 18 Μαΐου, αλλά το ερώτημα μου προς την Κομισιόν είναι τι θα γίνει μετά την αυριανή μέρα, εάν δεν έχουν να υπάρξει άλλα αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα. Θα επαναλάβετε αυτά που είπατε στην επιστολή σας που στείλατε στο Μπαγκλαντές πριν από δύο μήνες. Ο κύριος Καρίμ από το ECR για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να σας πω πάντα είναι χαρά για μας το να σας βλέπουμε στην Ολομέλεια. Και χαιρετίζω τον πολύ ανοιχτό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα εμπορικά θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαιρόμαστε και για τη διαφάνεια που μας προσφέρετε. Συνάδελφοι, τον Μπαγκλαντές λοιπόν. Το Μπαγκλαντές ε, είναι μια ιστορία, ένα νόμισμα με δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι αυτή για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο κυρίως μπορεί να νιώθει μεγάλη υπερηφάνεια. Παίξαμε ρόλο στο να υπάρξει ανάπτυξη. Διασφαλίσαμε το ότι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι της κοινωνίας του Μπαγκλαντές σήμερα βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου μπορούν να προσπορίζονται με υπερηφάνεια, με αξιοπρέπεια. Ε, το Κοινοβούλιο έχει επενδύσει σε όλα αυτά. Βλέποντας λοιπόν τα ουσιαστικά επιτεύγματα ε, αυτό είναι το ένα. Πρέπει όμως να δούμε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Και μου είναι απόλυτα σαφές ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές είτε δεν ακούει, ή επιλέγει να μην ακούει ή και δεν καταλαβαίνει το τι ακριβώς λέμε. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο επιθυμώ να εκπέμψω ένα σαφέστατο μήνυμα. Δεν έχει αυτό να κάνει με λεπτομέρειες. Κομισιόν ασχολείται με τις λεπτομέρειες. Εγώ θέλω απλά να πω στον Μπαγκλαντές ότι δεν θέλω κι εγώ και όλοι μας να υπάρξει μια κατάσταση όπου από τα χειροκροτήματα και τις επιθυμίες ε, για τη νίκη και τα ε, ουσιαστικά επιτεύγματα καταλήγουμε σε αρνητικά αποτελέσματα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να παραμείνουν οι πόρτες ανοιχτές για εσάς. Παρακαλώ λοιπόν λάβετε αυτό το μήνυμα, αντιδράσετε θετικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι της πρόοδου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σάντσες, η κυρία με συγχωρείτε Σάντσες, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Όντω, εδώ και τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια ε, σημειώθηκαν που τώρα να Πλάσα και οι εργαζόμενοι του Μπαγκλατές, κυρίως στο κλωστοϊφαντουργικό τομέα, έζησαν μια δραματική στιγμή αν και ορισμένοι μας παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα. Η ελευθερία της ε, έκφρασης, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν υπάρχουν στο Μαγκλατές. Και υπάρχουν πάρα πολλές αφαίρετες απόπειρες, εκβιασμοί, βασανιστήρια ε, συνδικαλιστών ε, και ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί η Κομισιόν, παρότι με ευχαριστούν τα όσα είπε η Επίτροπος εδώ, δεν πρέπει να κοφεύει. Θα πρέπει να ξεκινήσει μία έρευνη για έρευνα για παραβίαση διεθνών συμβάσεων για τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση, βλέπουμε ανησυχία ότι διάφορε πρωτοβουλίε εθελοντικέ για την βιωσιμότητα του ε, κλωστοφαντουργικού τομέα δεν λειτουργούν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν ε, να καταφέρουν να σταματήσουν οι, παραβία, οι παραβιάσει. Πριν από 15, 15 ευρωβουλευτέ ζητήσαμε. Α, να γίνει κάτι ε, στον κλωστοϊβαντουργικό τομέα. Σας παρακαλώ, ε, το, το έχουμε ζητήσει εδώ και μέρες αυτό το πράγμα. Κάντε κάτι. Ευχαριστούμε κυρία Σάντζες που μίλησε εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Τώρα η κυρία Χάουταλα από τους Πράσινους. Παρακαλώ Χάιντι, ένα λεπτό έχεις. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, σας ευχόμαστε καλή δύναμη αύριο στο Συμβουλίο που θα συζητήσει το θέμα της πρόοδου δηλαδή στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε το Μπαγκλαντές. Έχουμε σειρά ετοιμάτων ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Επίτροπε, συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που δεν διαπιστωθεί αισθητή πρόοδος στη συμμόρφωση, ότι υπάρχει ακόμα και σήμερα η προπτική να αποταθείτε στον Διεθνή Οργανισμό εργασία για να καταγγείλει τι παραβιάσει τη εργασιακή νομοθεσία. Διότι εν τέλει πρέπει να λάβουμε υπόψη μα σοβαρά αυτό το σύμφωνο βιωσιμότητα. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αλλάξουμε τι ζωέ αυτών των ανθρώπων. Αν όμως ε, η άλλη πλευρά δεν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, πρέπει να συναγάγουμε τις συμπεράσματά μα και να κάνουμε κάτι. Δεύτερον, Θυμίζω ότι 500 βουλευτές ζήτησαν ε, συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα πρώτη εργασίας. Να επαναλάβουμε αυτό το αίτημα είναι κάτι το οποίο απαιτείται για να ισχύσουν οι κανόνες ισότιμα για όλους. Ένα λεπτό για τον κύριο Τσόκα από το ΙΕΝΕΦ. Την ε, εβδομάδα που ο Τζαν Λούκα Μπονάνο έχει τα γενέθλιά του, θέλω να χρησιμοποιήσω και εγώ την, τον, τρόπο που επικοινωνεί ο Τζαν Λούκα. Αυτοί που κοιμάστε εδώ στην Ευρώπη, σας παρακαλώ να ανοίξετε τα μάτια. Ανοίξτε τα μάτια. Ξυπνήστε. Ξυπνήστε. Μην γίνεστε λακέδες των πολυεθνικών. Οι πολυεθνικές οι οποίες έδειξαν με τη στενοχή της Ευρώπης ότι μπορούν να σκοτώσουν την Ιταλία, όχι μόνο, ε, και σκότωσαν στην Ιταλία τον θαυμάσιο τομέα των κλωστοϊφαντουργικών. Αυτέ οι πολυεθνικέ, οι οποίε πάνε και παράγουν σε άλλε χώρε και που κερδοσκοπούν με καταστάσεις που τις βλέπουν όλες. Ε, χρησιμοποιώντας ανθρώπους ως σκλάβους, ε, χρησιμοποιώντας παιδιά ανήλικα που δουλεύουν 12, 13, 14 ώρες την ημέρα με 2 ευρώ τη μέρα χωρίς καμία προστασία στην, στο χώρο εργασίας. Είναι απαράδεκτο. Αν η Ευρώπη δεν θέλει να συνεχίσει να είναι συνένοχος αυτός των, αυτών των πολυεθνικών και αν δεν θέλει να είναι συνένοχη για αυτούς τους πολυάριθμους θανάτους στο χώρο εργασίας θα πρέπει και το τονίζω να σταματήσει αυτά τα παράνομα προϊόντα να, να μπαίνουν στην Ευρώπη. Ε, παράνομα προϊόντα που παράγονται χωρίς να σέβονται τους κανόνες. Οι, εργαζόμε, οι εργοδότες που παράγουν τέτοια προϊόντα ε, χωρίς να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι, παράγουν παράνομα προϊόντα. Ο κύριος Ζένφελτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι κρίμα που τραγωδίες είναι αυτοί του Μπαγκλητές πολλές φορές οδηγούν έστω και έτσι στην αλλαγή στον δρόμο δηλαδή της συμμόρφωσης με τους κανόνες και τα πρότυπα των δικαιωμάτων του ανθρώπου τις συνθήκες εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας κλπ. Η συμφωνία του Μπαγκλαντές με Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείε και τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας ε, βελτίωσαν την κατάσταση. Θεσπίστηκαν αλλαγές από το 2001 στην εργασιακή νομοθεσία. Περίπου 500 εγκαταστάσεις υποβλήθηκαν σε έλεγχο, δημιουργήθηκαν νέα συνδικάτα. τα οποία αναγνωρίστηκαν και επισήμω. Δημιουργήθηκαν νέοι θεσμοί. Όλα αυτά είναι θερικές εξελίξεις. Χάρη και στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του συμφώνου που δημιουργεί υποχρεώσεις για τις ίδιες επιχειρήσεις. Θα λέω ότι η πορεία αυτή είναι ακόμη εξελίξη, δεν φτάσαμε στον τελικό μας στόχο. Ας μην ξεχνούμε επίσης ότι σε χώρες όπως το Μπαγκλαντές οι επιχειρήσεις της περιοχής είναι μια λύση κατά της πίνες, της ενεργείας. Θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσεις, αλλά τις υλοποιήσουμε με τρόπο υπεύθυνο για να βοηθήσουμε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους στις πιο φτωχές χώρες χωρίς να καταδικάσουμε βεβαίως σε κατάρρευση και τις επιχειρήσεις, την βιομηχανία δηλαδή που δημιουργεί ευκαιρίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που παρακολουθείτε αυτό το θέμα. Ε, είναι σαφές ότι όσον αφορά τον Μπαγκλατές, ένα μεγάλο θέμα είναι η πρόσβαση στην αγορά. Και βεβαίω χαιρετώ το γεγονό ότι δεκάδε χιλιάδε εργαζομένων, κυρίω οι γυναίκε, ε, ε, ζουν, προσπορίζονται, βιοπορίζονται μάλλον από το άνοιγμα τη αγορά. Μα μας μίλησαν μάλλον οι γυναίκε όταν πήγαμε στον Μπαγκλαντέ για τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν και γι' αυτό και εμείς χαιρετίζουμε αυτά το που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Η επιστολή που στείλατε ε, ε, στον πρέσβη και αυτό ήταν ε, ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι καθαρά τεχνική αλλά περιλαμβάνει και τον σεβασμό για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, ένα θέμα που προκύπτει συνεχώς στο Μπαγκλαντές είναι το κατά πόσον οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές ε, όπου ισχύουν οι ίδιες και χειρότερες συνθήκες από ό,τι στο Μπαγκλαντές. Εσείς λοιπόν τι εγγύησεις ε, μπορείτε να μας δώσετε έτσι ώστε πράγματι να τηρούνται οι κανόνες του ILO και τα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, ευθύνη που φέρουν οι εταιρείε μας, δεν είναι δυνατόν να γίνονται επενδύσεις αν και οι άνθρωποι δεν έχουν αξιοπρεπείς και καλές τιμές τιμές για τα προϊόντα που παράγουν. Είχαμε μια σχετική έκθεση τον προηγούμενο μήνα και Τώρα η Κομισιόν χαιρετίζει, ε, παρουσιάζει μια λυσίδα ε, της αξίας έτσι ώστε να καταβάλλονται οι σωστές τιμές για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στο Μπαγκλαντές, ε, κυρίως τα κλώστο υφαντουργικά. Ο κύριος Λάμπερτ, η κυρία Λάμπερτ, με συγχωρείτε, Ευχαριστώ και εγώ για το ενδιαφέρον τη Επιτρόπου στον τομέα του έτοιμου ενδύματο στο Παγκλαδέσιο αλλά και αλλού. Και εδώ ομιλώ ω πρόεδρο της Ενπροσωπεία για την Νοτιοανατολική Ασία. Παρακολουθούμε το Σύμφωνο Βιωσιμότητα από την αρχή και πρέπει να σας πω ότι από πολλούς θεωρείται μια καινοτόμος ανταπόκριση Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τραγικά γεγονότα του Ραναπλάζα. Πλάζα. Είναι ίσω και μοντέλο πρότυπο θα έλεγα για την εμπλοκή μα σε άλλε χώρες. Η κυρία Μακάβαν έχει δίκιο ότι το Μπαγκλαντέ δεν είναι η μόνη χώρα με προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι πολλοί μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα για την βελτίωση των σχέσεων με τον Μπαγκλαντέ και την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Θέλουμε όμω η πορεία αυτή να συνεχιστεί, να ανανεωθεί, να ενισχυθεί. Γιατί αυτό θα είναι και η ευκαιρία για τον Μπάγκλαντες να αποδειχθεί ηγέτης. Ηγέτης όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο, τα συνδικάτα, την υπεύθυνη παραγωγή. Όπως και εμείς βεβαίως πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, να εξασφαλίσουμε μια αλυσίδα εφοδιασμού χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο για ένα λεπτό. Πήγα το Μάρτι στο Μπαγκλαντές με την αντιπροσωπεία της πολιτικής ομάδας. Και έτσι είδατε ότι συμβαίνει. Ε, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε κάποια βελτίωση τουλάχιστον στα εργοστάσια που κατασκευάζουν παπούτσια. Ε, είχαν πρόσφατα ε, συλληφθεί οι συνδικαλιστές. Ε, βεβαίως ισχύει το ότι εξακολουθούν να παραβιάζουν σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα και οι προδιαγραφές. Εμεί ζητήσαμε να υπάρξει βελτίωση και ως εκ τούτου ε, έχουμε αυτή την ανακοίνωση κομισιών ε, που είναι πολύ σημαντική. Ε, περιμένω να δω τι θα γίνει με αυτό το σύμφωνο της βιωσιμότητα και με ενδιαφέρει κυρίως το τι θα κάνει η Κομισιόν έτσι ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το σύμφωνο βιωσιμότητας. Σας παραπέμπω Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση πρωτοβουλία του Απριλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αλυσίδα τροφοδοσίας στην κλώστο εφαντουργία. Ε, το Κοινοβούλιο ζητάει από την Κομισιόν νομοθετική πρόταση που επιτέλους ε, θα επιβάλλει και θα ζητάει το να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές σε αυτή την αλυσίδα τροφοδοσίας. Γιατί νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες συμπεριλαμβανομένου και του Μπαγκλαντές. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λίτσο και τώρα στο κάτσο. Ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ ένα λεπτό. Grazie, Presidente. Έχουμε επανειλημμένα ασχοληθεί με την εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί στο Μπαγκλαντές. Εκεί όπου εργάζονται μικρά παιδιά 10 και 12 ώρες εκεί όπου παραβιάζεται βάναυσα η εργασιακή νομοθεσία εκεί όπου έχουν καεί ζωντανοί εκατοντάδες εργαζόμενοι στη ράνα πλάζα εκεί όπου οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές αφού έκλεισαν τις υφαντουργίες στην ευρώπη έκτισαν εργοστάσια όπου δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι για ένα κομμάτι ψωμί. δεν πρόκειται το μπαγκλαντές να συμμορφωθεί να είστε σίγουροι. θα μας κοροϊδεύει και η κυβέρνηση του μπαγκλαντές και οι πολυεθνικές. θα παίζουν το κρυφτούλι μόνη λύση η απαγόρευση εισαγωγής ενδυμάτων και άλλων κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων από τον μπαγκλαντές λήψη μέτρων για την αναβίωση της ευρωπαϊκής κλωστοϊφαντουργίας με παροχή ειδικού καθεστώτος για τον κλάδο αυτό τόσο στην ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου. ευχαριστώ. pozorně Κύριε Επίτροπε, με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ε, θέλετε να αγωνιστείτε για εκείνους ε, οι οποίοι αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς πιστεύουμε ότι ε, είναι σημαντικό να ε, περασπίζεται κανείς τα δικαιώματα όπως και την ελευθερία της ε, άποψης και του συνεταιρίζεστε. Πολύ σημαντικό το ότι ασχολούμεθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το εργασιακό δίκαιο στο Μπαγκλαντές. Εγώ έχω μελετήσει τα διάφορα κείμενα και τώρα είμαι πολύ επιφυλακτική όταν αναφέρεται ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές είναι πρόθυμη να λάβει υπόψη της το ψήφισμα και να βελτιώσει την κατάσταση. Ελπίζω λοιπόν λοιπόν αύριο κάτι να γίνει και αν δεν γίνει κάτι μέχρι τις 18 Μαΐου ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα έτσι ώστε να μην έχουμε πλέον να κάνουμε με ε, διπλωματικές πομφόλιγες. Η κυρία Μάλμστρομ για την απάντησή της. Ευχαριστώ όλους. Πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση συμμερίζομαι τους ε, στόχους που θέλετε και εσείς θα κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε. Και θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα στην επικοινωνία μας με τον Μπαγκλαντές. Γιατί θέλουμε οι σύνδικες εργασίας να είναι εξωπερπείς. Το Σύμφωνο Βιωσιμότητας είναι, όπως είπατε και πολλοί από εσά, ε, πρακτικά μοναδικό. Είχε ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να ενημερωθούν, συμμετέχουν εκεί η κοινωνία των πολιτών, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι. Έχουν γίνει πολλά. Όχι αρκετά, αλλά κάτι έχει γίνει. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν, δεν ενδιαφέρονται, να αρχίζουν να ενδιαφέρονται. Κάτι κάνουν, δείχνουν εταιρική υπευθυνότητα, συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις, τουλάχιστον δέχονται επιθεωρήσεις από ανεξάρτητους φορείς. Και έτσι η παραγωγή τους γίνεται πιο αηφορική. Έγιναν πολλά λοιπόν. Υπάρχει πρόοδος, αλλά επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, δεν είναι αρκετή. Η κυβέρνηση λοιπόν του Μπαγκλαντές πρέπει να κάνει και άλλα. Πρέπει να κάνει, θα έλεγα, πολύ περισσότερα. Αύριο Έχουμε μια συνάντηση με τις αρχές του Μπαγκλαντές. Θα δούμε τι σκοπεύουν να κάνουν, τι κάνουν, αν έχουν μια στρατηγική, τη στρατηγική που ζητήσαμε και θα τα συζητήσουμε όλα σε κλίμα φιλικό και ειλικρινές. Αν κάτι πάει καλά, υπάρχουν προφανώς μέτρα τα οποία θα λάβουμε και θα τα λάβουμε, όχι μόνο σήμερα. Η συνάντηση είναι αύριο, ας τους δώσουμε μια ευκαιρία να μας δείξουν τι προτίθεται να κάνουν και φυσικά έχουμε και άλλα μέτρα πίεση. Το καταστήσαμε σαφέ στο Μαγκλαντέ ότι οι τέσσερι συστάσει του ILO, του Διεθνού Οργανισμού Εργασία, για παράδειγμα για την τροποποίηση τη εργασιακή νομοθεσία για να είναι σε συμμορφώση με τη συμβάση του ILO. Δεύτερον, ο νόμο για τι ελευθερέ ζώνε εξαγωγών επιτρέπουν 100% την ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Τρίτον, όλε οι πράξει έχουν γίνει κατά συνδικαλιστών να διερευνηθούν, να γίνουν σχετικέ ανακρίσει και τέταρτον οι αιτήσει καταχώρηση συνδικάτων να γίνονται μέσω αποδεκτές ε, εκτό βεβαίω αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι οι τέσσερι πιο σημαντικέ και κατεπίγουσε συστάσει μα. Αυτά θα τα ζήσουμε αύριο. Όσον αφορά τώρα τον οικονομικό και νομικό έλεγχο ορισμένων συμφωνιών, ε, το πράγμα δεν είναι πολύ απλό στον τομέα του ετοιμού ενδύματος. Συνεργαζόμαστε και με τον ΑΕΛΟ και με τον ΟΣΑ για να υλοποιηθεί στην πράξη, υλοποιηθούν στην πράξη αυτή η έλεγχη ε, και να βεβαιωθούμε ότι ακολουθούν στην, σε καθημερινή βάση. Είναι πάρα πολύ το, το πράγμα. Εμπλέκονται πάρα πολλές επιχειρήσεις και άλλοι συμμετέχοντες, αλλά εμπλεκόμενοι. Ήδη υπάρχει νομοθεσία για την εταιρική υπευθυνότητα και για την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά. Ε, έχουμε την οδηγία για την δημοσιοποίηση στοιχείων για κάποιες μεγάλες εταιρείε που ισχύουν και για τον τομέα του έτοιμου ενδύματος. Και επίσης συνεργαζόμαστε με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και με άλλους εταίρους στην περιοχή με στόχο να υποστηρίξουμε την αλλαγή, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να τον ενθαρρύνουμε και εν τέλει να οργανώσουμε και συναντήσεις με όλους τους εμπλεκομένους ώστε να υπάρχει συμμετοχή και πρόοδος πολιτική και οικονομική. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν, προσβλέπω σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο από εδώ και πέρα και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για να γίνουν θετικέ αλλαγέ για του εργαζόμενου, για τα συνδικάτα και εν τέλει για τον κόσμο, για τον πληθυσμό στον Παγκλαντέ, κυρίω γυναίκε και παιδιά. Μα χρειάζονται και πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε εκεί και ότι αγωνιζόμαστε. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σα, τη συζήτηση και τι προσπαθίε σα. Θα επανέλθουμε βεβαίω στο θέμα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο Μάλστρομ που ήρθε εδώ για να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Κλείνει η συζήτηση. Η ψηφοφορία για το ψήφισμα θα γίνει τον Ιούνιο. Και τώρα